Η Πρόεδρος, συνάδελφε, αρχίζουμε την συνεδρίαση. Θα ακούσατε ότι η δουλειά μας ε, τώρα είναι η συνέχεια της προηγούμενης δουλειάς μας όσον αφορά τις συζητήσεις μας δηλαδή για το μέλλον της Ευρώπης. Η δημοσία ακρόαση όσον αφορά τις δογματικές πτυχές ε, της κοινωνικής διάστασης της ε, Ένωσης. Είναι θέμα που το έχουμε συζητήσει, το έχουμε θεωρήσει πολύ ε, σημαντικό θέμα και, και θέμα ουσιαστικής σημασίας την τελευταία διετία συχνά έχει γίνει μια τέτοια συζήτηση σε σχέση με την λειτουργία της Ένωσης και επίσης στα πλαίσια της ε, κρίσης την οποία περάσαμε πριν από μία δεκαετία. Είναι επομένω πολύ σημαντική η ακρόαση. Και γίνεται στα πλαίσια της ε, έκθεσης από την Μπάρμπαρα Σπινέλη της Γκούε και ο κύριος Καστάλντο του EFTD ως συνεισήγητες. Και το θέμα σχετίζεται και με τις ε, ευρωεκλογέ που θα γίνουν του χρόνου. Είναι θέμα επαφής μας με τον κόσμο. Γι' αυτό και σας ευχαριστούμε που ήρθατε και θα σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο. Τώρα το ποιος θα αρχίσει βρείτε το μεταξύ σας. Ο κύριος Φαντενμπρούκε θα δώσει τον εκτήριο λάκτισμα και η κυρία θα έχει την τελευταία λέξη. Πολύ ωραία προσέγγιση. Έχετε το λόγο κύριε καθηγητά μεταδίδεται στο ίντερνετ το διαδίκτυο. Οπότε προσέχτε να είστε χαμογελαστή και να μην βρίζετε. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Στα 15 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου θα ήθελα να επικεντρωθώ σε αυτό που αποκαλώ εγώ ενοιολογική διευκρίνηση Κάτι που χρειαζόμαστε, πιστεύω, όταν συζητούμε την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπωσδήποτε σε μια επιτροπή σταγματικών υποθέσεων, όταν εξετάζουμε την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τους στόχους και τις πιθανές θεσμικές προεκτάσεις. E Θα ήθελα να ξεκινήσω από την ορολογία. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις, μελέτες, βιβλία που μιλούν για την κοινωνική Ευρώπη. Όμως πρόκειται και μια εξαιρετικά ασαφή διατύπωση. Για παράδειγμα, πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να βρει ε, τον όρο κοινωνική Γερμανία στη βιβλιογραφία. Ποτέ δεν ε, χρησιμοποιείται μια τέτοια διατύπωση. Όταν ε, μιλούμε για την κοινωνική πολιτική στη Γερμανία, λέμε ότι η Γερμανία είναι ένα κράτος πρόνοιας, ομοσπονδιακό κράτος, ε, έχει στόχους, αποστολές, έχει σύνταγμα και όλα αυτά τα στοιχεία τα παίρνουμε υπόψη κατά αυτή τη συζήτηση. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται να έχουμε μία γενική και αόριστη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να το εξετάσουμε λοιπόν από θεσμικής άποψης. Και αν ρωτήσετε τι εννοείται με την κοινωνική Ευρώπη, Κάποιοι θα απαντήσουν λιγότερη Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει σε πάρα πολλού τομεί. Άλλοι θα πούνε η κοινωνική Ευρώπη σημαίνει περισσότερη Ευρώπη. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει ε, και την αμφισημία αυτή τη έννοια. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούμε μια διαφορετική διατύπωση που μπορεί να μην είναι τόσο ελκυστική και δημοφιλής. Δεν πάω να πείσω τους ψηφοφόρους, για παράδειγμα, με αυτήν, αλλά διευκρινίζει και αποσαφηνίζει το διακύβευμα. Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ένωση. Εγώ έτσι την αποκαλώ, γιατί πρώτον ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας. Είναι μια ένωση εθνικών κοινωνικών κρατών. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, ένα περιβάλλον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άνθηση των εθνικών κρατών πρόνοιας. Για να το επιτύχουμε αυτό, και αυτό είναι και το πιο δύσκολο, για να δημιουργήσουμε λοιπόν αυτή την ένωση, ε, θα πρέπει να στηρίξουμε το εθνικό κράτος πρόνοιας στις συστημικές του λειτουργίες, όμως σε μερικές από αυτές τις λειτουργίες, όχι όλες. Θα σταθώ σε ένα παράδειγμα. Δίκαιη και αποτελεσματική εταιρική φορολογία στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όμως ίσως χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για να το πετύχουμε, για να στηρίξουμε αυτή την βασική λειτουργία. Δεν θέλω να επεκταθώ. Να πάω σε ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο γνωρίζω και καλύτερα, οικονομική και κοινωνική σταθεροποίηση. Το επιχείρημα μου εν είναι ότι αν θέλουμε μια πραγματική ένωση κρατών πρόνοιας που υποστηρίζουν λοιπόν τα εθνικά κράτη πρόνοιας σε ορισμένες από τις βασικές τους λειτουργίες, προφανώς θα πρέπει να συμφωνήσουμε τα βασικά κριτήρια, τους βασικούς στόχους που θα κατευθύνουν τη δράση μας. Η Ένωση λοιπόν των κρατών πρόνοιας χρειάζεται γενικά κριτήρια και στόχους, αλλά χρειάζεται και μία βασική συνένεση για τους στόχους και τα πρότυπα που θα ισχύσουν, θα εφαρμοστούν. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, σημαίνει ότι οι χώρες θα έχουν συγκεκριμένο κοινωνικό στόχο στο πλαίσιο της Ένωσης, θα ε, προωθούν και την άνθηση των εθνικών κρατών πρόνοιας, αλλά και μια πανευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή. Μία σύγκληση προς τα πάνω με σκοπό την ευημερία. Είναι κάτι το καινοφανές και το πρωτότυπο? Όχι. Αυτό ήταν και το όραμα των ιδρυτών ε, του Ευρωπαϊκού εγχειρήματο που διαπραγματεύτηκαν ε, την ε, συνθήκη της Ρώμης το 1958. Ανοδική σύγκληση λοιπόν, άνθηση των κρατών πρόνοια. Αυτό αποτέλεσε την έμπνευση για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Εδώ λοιπόν δεν ξεκινάμε από την αρχή, θέλουμε απλώς να δούμε πώς ε, θα το μεταφέρουμε αυτό στην πράξη. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μεταφράζεται στην πράξη όλο αυτό το όραμα της ανωδικής ε, σύγκλησης. Γι' αυτό πρέπει να επανεξετάσουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να περάσω τώρα στο παράδειγμά μου για την ε, σταθεροποίηση. Για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Θα με, περάσω μετά εν συντομία και στην ε, εσωτερική αγορά των 27. Αλλά πρώτα για την ΟΝΕ. Και συγγνώμη για τις αξιωματικές μου θέσεις. Όλο ένα και περισσότερο να γνωρίζουμε ότι για να λειτουργήσει σωστά η ΟΝΕ πρέπει σε ένα βαθμό τουλάχιστον να συγκεντρώσουμε τη διαχείριση ορισμένων κινδύνων όπως η τραπεζική κίνδυνη. Χρειάζεται ένας βαθμός ε, συγκέντρωσης και διαχείρισης ε, των τραπεζικών κινδύνων. Δεν είναι εύκολο αυτό το θέμα, όμως σε μεγάλο βαθμό οι περισσότερες νομισματικές ενώσεις μιλούν και για την ε, ασφάλιση των ανέργων ε, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί αρχικά έχουμε την συγκέντρωση ε, των κινδύνων για να αντιμετωπίσουμε τους ασύμετρους κινδύνους έτσι υπάρχει ένας επιμερισμός και αν δείτε και την ιστορία των ΗΠΑ εξετάζουμε και την θετική εξωτερική διάσταση με την εύρυθμη λειτουργία των εθνικών σταθεροποιητικών μηχανισμών που είναι ζητήματα δημοσίου συμφέροντος ε, σε μια νομισματική ένωση. Είναι θετικό κάθε κράτος μέλος να έχει μια, ένα τέτοιο ε, μηχανισμό σταθεροποίησης. Αλλού μίλησα και για μια εμβολιαστική ε, δράση, αλλά δεν θα το κάνω εδώ. Αλλά αυξάνεται η εντύπωση και διαβίνεται αυτή η εντύπωση ότι αρχικά χρειαζόμαστε ένα τέτοιο μηχανισμό σταθεροποίηση στο ιστορικό των κρατών μελών και για την ανεργία και του κραδασμού που συνδέονται με αυτήν. Και μετά, ακολουθώντας αυτή την άγουσα, χρειαζόμαστε, για παράδειγμα, ένα επαρκώς ε, γενναιόδωρο σύστημα ε, επιδομάτων ανεργία, καλή κάλυψη, να μην υπάρχει καταγερματισμό τη αγορα εργασίας που οδηγεί σε πολύ κακή ασφάλιση ε, ορισμένου τμήματος ε, του ανθρώπινου δυναμικού, να μην προάγονται ε, εργασιακές σχέσεις που δεν εντάσσονται στην κοινωνική ασφάλιση, να δραστηριοποιηθούν οι άνεργοι και να έχουμε και κατάλληλες ζώνες προστασίας και μηχανισμούς προστασίας. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να υλοποιηθούν για να έχουμε έναν καλό μηχανισμό σταθεροποίησης σε όλα τα μέλη. Αυτό θα ήταν το καλύτερο αν θέλαμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, μία τέτοια ρύθμιση. Δεν θέλουμε δηλαδή να έχουμε επιμερισμό κινδύνων σε μια ομάδα κρατών, από τις οποίες κάποιες ε, δείχνουν ιδιαίτερη προσήλωση στο μηχανισμό σταθεροποίησης και βλέπουν ότι λειτουργεί καλά, ενώ άλλες όχι. Και λένε εντάξει, απλώς θα μας καλύψει. Χρειαζόμαστε λοιπόν κοινού κανόνες και πρότυπα για την ποιότητα των εθνικών συστημάτων σταθεροποίησης. Αν σκεφτείτε για ένα μέλλον όπου μπορεί να υπάρξει επιμερισμός ε, των κινδύνων σε ενωσιακό επίπεδο. Να το διευρύνουμε τώρα λίγο. Αν σκεφτείτε την κοινωνική διάσταση μίας ε, νομισματικής ένωσης, από λειτουργική άποψη, άποψης, ποια είναι η κοινωνική διάσταση που προκύπτει από την ΟΝΕ, που δεν ήταν αυτό που είχαν κατά νου οι ιδρυτές. Τώρα όμως έχουμε νομισματική ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια κοινή αντίληψη της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό σε μια ΟΝΕ. Ναι. Χρειαζόμαστε θεσμούς της αγοράς εργασίας ε, που μπορούν να οδηγήσουν σε συντονισμό των μισθών για να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα. Και τώρα κάτι το οποίο προκύπτει ε, αντικειμενικά από την επιστημονική έρευνα Για να γίνει αυτό απαιτούνται οι συλλογικέ εμβάσει εργασία. Παντού. Αυτό δεν είναι προσωπική μου γνώμη. Και μετά χρειαζόμαστε και έναν ε, πυρήνα ε, πολιτικών αρχών που ενθαρρύνουν και προάγουν την ικανότητα σταθεροποίηση των πρώτων μελών, αλλά αποτελούν και προϋποθέσεις για το μέλλον, όπου θέλουμε να περάσουμε σε ενωσιακό επιμερισμό κινδύνων. Είναι μικρός αυτός ο κατάλογος, αλλά αποτελεί μια βάση κοινών προτύπων. Και δεν είναι τυχαίο ότι θα βρείτε αυτές τις αρχές, όχι με την ακριβή διατύπωση, αλλά αρκετά κοντά στον ε, Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που δημοσιεύτηκε πέρσι. Κάτι που προετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη έχοντας ακριβώς κατά νου την προβληματική της ΟΝΕ. Ναι, κατά ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά εξηγούνται με μια σωστή και ορθή δυνατότητα και ικανότητα σταθεροποίηση. Επιστρέφουμε μέσω αυτού στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Οι ιδρυτέ λοιπόν ε, δεν το είχαν σκεφτεί, γιατί δεν υπήρχε και η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Κλείνοντα, Δύο λόγια για την Ένωση των 27 και την εσωτερική αγορά. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε, δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά ε, τα γνωρίζετε κι εσείς, Ποιε είναι οι διαφορέ μεταξύ του 1958 και του 2018. Είχαμε τότε έξι χώρε, παρόμοιε μεταξύ του συγκρίσιμε ε, σε, από πλευρά ανάπτυξης ε, και δομής του κράτου πρόνοια. Τώρα έχουμε 28 από το χρόνο 27 με πολύ μεγάλες ανομοιογένειες και δομές ε, στο κράτος πρόνοιας. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανομοιογένεια ε, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο. για να έχουμε το κανονιστικό πλαίσιο της δίκαιης κινητικότητας ε, Πολλοί εργάζονται από αυτού. Πρέπει να διατηρήσουμε την αρχή της ελεύθερης ε, κυκλοφορίας. Υπάρχει βέβαια και η εξαίρεση της απόσπασης εργαζομένων. Εγώ, εν είδη παραδείγματος, θα έλεγα ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο χρειαζόμαστε ένα καθεστώς διασφάλισης του κατώτατου μισθού. Όχι του ενιαίου κατώτατου μισθού, γιατί αυτό είναι μια ανοησία, αλλά ε, καθολικές αρχές ε, του καθεστώτος του κατώτατου μισθού. Για να είναι αυτό το καθεστώς προβλέψιμο και διαφανές, για να μπορεί και η εστρική αγορά να λειτουργεί σωστά. Και πάλι θα βρείτε ορισμένα ψήγματα αυτής της αντίληψης και στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Δεν ε, εφευρίσκουμε εκ νέου λοιπόν τον τροχό εδώ. Οι ιδρυτές είπαν ότι θεωρούσαν ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα οδηγήσει σε σύγκληση προς τα πάνω και ευημερία. Αυτή είναι η έμπνευση που διατηρούμε και σήμερα. Όμως πρέπει να επανεξετάσουμε την αγορά εργασίας, την ένωση των κρατών πρόνοιας που θα δημιουργήσει μια νέα κοινωνική ένωση, θα επιτρέπει στα κράτη πρόνοιας να ανθίσουν και να ευημερήσουν, Χρειάζεται μια συγκέντρωση της διαχείρισης κινδύνων, αυτόματος μηχανισμού σταθεροποίησης. Αυτό αναπόφευκτα ε, προϋποθέτει και συνένεση σε μια σειρά κοινωνικών προτύπων. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο εύρυθμης λειτουργίας στην ε, Ένωση των 27 και αυτό προϋποθέτει κοινωνικά πρότυπα. Δεν θα παρουσιάσω την επόμενη διαφάνεια γιατί θα τα πει και συνάδελφος στη συνέχεια. Αφορούσε ακριβώ ε, τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και πώ μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Με δύο λόγια λοιπόν, για να μην ξεπεράσω το χρόνο μου. Δεν χρειάζεται τροποποίηση τη συνθήκη για να έχουμε αποτελέσματα στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Έχουμε επαρκή μέσα τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο και μάλιστα με συμπληρωματικό τρόπο. Έχουμε μία σειρά νομικών μέσων. Έχουμε τα ευρωπαϊκά ταμεία και έχουμε και κάτι πολύ σημαντικό, το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Τώρα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα μέσα για να έχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Δεν χρειάζεται νέα συνθήκη. Υπάρχει συζήτηση κατά πόσο κάποια στιγμή θα έχουμε αυτόματους δημοσιονομικούς σταθεροποιητές και αν όλα αυτά θα συνδέονται με κραδασμούς στην αγορά εργασίας. Και όλο αυτό συνδέεται με την αντασφάλιση των ανέργων. Αν απαιτείται τώρα τροποποίηση της συνθήκης, μπορώ να σας στείλω και στοιχεία, η απάντηση είναι όχι. Είναι μεγάλη συζήτηση βέβαια. Θα μιλήσει και ο επόμενος ομιλητής για αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται να μας απασχολήσει μια τέτοια τροποποίηση της συνθήκης. Ήδη με τα εφιστάμενα μέσα μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τώρα λίγο διαφήμιση, το ξέρω, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι και χρήσιμο μαζί με την Κάθριν ε, Μπάρναρτ και τον Χέρτε Τεμπάρε, που είναι ερευνητής. Έχουμε δημοσιεύσει, έχουμε κάνει αυτές τις δημοσιεύσεις για την ε, αρχή της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ένωσης. Θα βρείτε το πρώτο κεφάλαιο στο Open, σε ανοιχτή μορφή, στο διαδίκτυο, αλλά αν σας ενδιαφέρει υπάρχει και το τρίτο τμήμα Εκεί ο Κουν Λέναρτς, πρόεδρος του δικαστηρίου όπως γνωρίζετε, μιλάει για τον τρόπο που μπορεί να αξιοποιηθεί η συνθήκη για την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης. Και τι σημαίνει αυτό. Ένα κεφάλαιο λοιπόν που κοιτάζει και εξετάζει ανάντι αυτή τη θεσμική διαδικασία. Τα κράτη-μέλη δηλαδή τι θεωρούν ε, από, από άποψης τα πιο σημαντικά στοιχεία. Και μετά έχουμε και δύο κεφάλαια που μελετούν τα, τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες ε, της Ένωσης και του νομοθετικού μας πλαισίου. Υπάρχουν πολλοί πόροι, πολλά στοιχεία στο σημερινό ευρωπαϊκό συνταγματικό πλαίσιο. Και εντάξει, οι ειδικοί μπορεί να μας πούνε πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, αλλά έχουμε πολλά μέσα στη διάθεσή μας, αρκεί να έχουμε σαφείς στόχους. Να γνωρίζουμε πραγματικά γιατί θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατών Πρόνοιας. Τι ενέχει αυτή η υπερεθνική πρωτοβουλία. Κλείνοντας, μία μικρή επίκριση. Είναι λίγο άδικο γιατί δεν είναι εδώ οι εισηγητές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει δημοσιεύσει ένα έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση εγώ είμαι μάλλον επιφυλακτικό, Παρουσιάζει ενδιαφέρον βέβαια, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και μία εσφαλμένη αντίληψη σε αυτό το έγγραφο. Ότι μπορούμε να έχουμε ό,τι θέλουμε σε οποιαδήποτε μορφή. Ότι μία ομάδα κρατών μελών κάνει το α σε έναν κοινωνικό τομέα, ένα άλλο σύνολο κρατών κάνει το β με διαφορετική δομή, ένα τέτοιο μοσαϊκό ας πούμε. Εγώ δεν συμφωνώ. Αν θέλουμε να προσθέσουμε μία κοινωνική διάσταση στην ΟΝΕ, ναι, αυτό αφορά όλα τα κράτη που συμμετέχουν στην Νομισματική Ένωση, όχι για ορισμένα. Και για την εσωτερική αγορά, αν θέλουμε να σαγάγουμε συγκεκριμένα μέσα, το μισθό και το καθεξής. Αυτό είναι ένα πλαίσιο για όλους. Θα μπορούσαμε ε, να διαφοροποιήσουμε λίγο τα πράγματα μεταξύ ΟΝΕ ναι και εσωτερική αγορά για να δούμε πώ θα αναπτυχθούν τα πράγματα σε ενωσιακό επίπεδο. Αλλά κατά τα λοιπά δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο διαφοροποίηση. Οι κοινωνικές πολιτικές που εξετάζουμε τώρα είναι θέμα δημόσιας τάξης, δημόσιας ένομης τάξης που δημιουργείται πλέον. Οπότε δεν με ικανοποίησε πολύ η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Και στην τρίτη δημοσίευση που αναφέρω έχω παραθέτω ορισμένα επιχειρήματα. Λοιπόν, δεν μπήκα στα πραγματικά νομικά ζητήματα, αλλά αν, μπορείτε, αν θέλετε μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον ε, Φρανσίσκο Κωνσταμάνη. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε σήμερα εδώ και είναι τιμή μου που βρίσκομαι στη σημερινή ακρόαση. και η δική μου παρέμβαση εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, επειδή έχουμε βέβαια και συγκεκριμένο χρονικό περιορισμό κατά την παρέμβασή μας. Ε, εστιάζω λοιπόν ε, στη σχέση ανάμεσα στο οικονομικό και το κοινωνικό σχέλος ε, της Ευρωπαϊκής Δικασίας Ολοκλήρωσης και θα εστιάσω ιδιαίτερα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. και εδώ ε, και στα όσα είπε μόλι τώρα ο καθηγητή Βαντεμπρούκε, ε, τονίζω ότι πριν από οποιαδήποτε μεταρρύθμιση τη συνθήκη θα πρέπει να διασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή στο ακέραιο των υφιστάμενων συνθήκων. Γιατί η δική μου αίσθηση, και δεν είναι απλώ και μόνο αίσθηση, είναι ότι η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση λειτουργεί με τρόπο τέτοιο τη σήμερα ημέρα που δεν ευθυγραμμίζεται πλήρω με τη συνθήκη και με το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων μία από τις ε, πιο εμ, ορατές αν θέλετε εξελίξεις που παρατηρήσαμε για την τελευταία δεκαετία ήταν το γεγονός ότι η η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποτάχθηκε, ως κοινωνική στόχη δηλαδή, στους οικονομικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο οδήγησε βέβαια και στη διάβρωση της νομιμότητας της όλης διαδικασίας ολοκλήρωσης. Ε, άρα λοιπόν κατά το πρώτο τμήμα της ε, παρουσίασής μου θα κάνω ένα βήμα προς τα πίσω για να ρίξω μια ματιά στο πώς τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι ώστε να δώσω το υπόβαθρο για το δεύτερο τμήμα της παρουσίασης όπου θα σας πω Ποια είναι η άποψή μου για το μέλλον. Ε, το έγγραφο λοιπόν που ε, συνέταξαν η Μπάρμπαρα Σπινέλη και ο Φάβιο Καστάλο τονίζει και συμφωνώ με, την, ε, αυτό το πόρισμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορισμένα περιθώρια δράσης στο κοινωνικό τομέα. Ωστόσο ένα στοιχείο που συχνά παραγνωρίζεται είναι το γεγονός ότι η επιλογή ε, του, τα κοινωνικά ζητήματα να παραμείνουν εκτός της εμβέλειας των υπερεθνικών ε, θεσμικών οργάνων ήταν μια επιλογή που έγινε προκειμένου τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να ασκούν τα δικά τους κοινωνικά ή να αναχαίρουν το δικό τους κοινωνικό προνομίο. Και με αυτόν τον συμβιβασμό μαζί με τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς ο στόχος ήταν να ενισχυθεί η αναδιανεμητική ικανότητα των ε, ε, εθνικών αρχών έτσι ώστε σε γενικές γραμμές να έχουμε μια αναβάθμιση ε, των κοινωνικών προτύπων. Αποφασίστηκε λοιπόν γενικά ότι δεν θα είναι αρμόδια τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινωνικά ζητήματα ακριβώς με στόχο την ανύψωση των κοινωνικών ε, προτύπων. Και de jure αυτή, αυτός ο συμβιβασμός συνεχίζει να ισχύει. Δηλαδή αν συγκρίνουμε τη συνθήκη, ε, τη συνθήκη της Ρώμης με τη συνθήκη της Λισαβόνας για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κοινωνικές διατάξεις δεν έχουν ε, τροποποιηθεί. Έχουν προσθεθεί νέες διατάξεις οι οποίες ενισχύουν ε, ακριβώς την εθνική κυριαρχία ε, των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα. Αν ρίξουμε για παράδειγμα μια ματιά στο άρθρο 9 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα διαπιστώσουμε ότι αναφέρει εκεί ότι τα, κράτη, τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσει που σχετίζονται με την ε, προώθηση ενός υψηλού επίπεδου απασχόλησης, ε, την ε, κατάλληλη κοινωνική προστασία, την καταπολέμηση του κοινωνικού απλουσμού, ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Αλλά αν τώρα πάμε από το de jure στο de facto, θα δούμε ότι αυτός ο αρχικός συμβιβασμός δεν ισχύει πλέον εδώ και καιρό. Και αυτό καθίσταται πιο σαφέ, ειδικότερα στο πλαίσιο τη νέα ε, οικονομική ε, και νομισματική ένωση, στο πλαίσιο δηλαδή τη νέα οικονομική διακυβέρνηση. Η, νέα λοιπόν διακυβέρνηση αυτή δίνει σε ορισμένα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια πρωτόγνωρη ε, δυνατότητα, εξουσίες δηλαδή σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό αλλά και την εποπτεία και την καθοδήγηση της πολιτικής σε τομείς οι οποίοι είναι ε, Εθνική αρμοδιότητας όπως για παράδειγμα οι μισθοί, οι συντάξεις, διατάξει ε, ε, απόλυσης και ούτω καθεξής. Και το βασικό πρόβλημα κατά τη δική μου άποψη είναι ότι αυτοί, αυτές οι εξουσίες εξυπηρετούν την επιτεύξη των στόχων της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης όχι κοινωνικούς στόχους όπως για παράδειγμα η αξιοπρέπεια, η αυτονομία, η κοινωνική δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν η κοινωνική διάσταση έχει μεταβληθεί σε μια ε, μεταβλητή, αν θέλετε, προσαρμογή, η οποία είτε θα πρέπει να μειώνεται προκειμένου να ε, μειωθεί ο σχετικό προπολογισμό του κράτους μέλου ή θα πρέπει να ε, συμβάλλει στην βελτίωση τη εξωτερική ανταγωνιστικότητα του κάθε κράτους μέλου. Άρα λοιπόν αυτή η μεταβολή, αν θέλετε αυτή η μετάλλαξη, ε, στην περίπτωση του εξαμήνου ειδικότερα, έχει, δημιουργήσει, έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός υβριδικού πλαισίου, ε, το οποίο επιτρέπει το συντονισμό και την ε, εποπτεία από την Επιτροπή σε μια σειρά από διαφορετικούς τομείς, έχοντα έτσι δυνατότητα να ασκεί πιέσει σε ό,τι αφορά τέτοιου είδου διαδικασίε, με την απειλή αυστηρών κυρώσεων. Και στην περίπτωση των πακέτων διάσωση, αυτό έχει γίνει ξεφεύγοντα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και τη λογική τη και τι εγγυήσει τη. Έτσι ώστε δηλαδή να αξιοποιηθεί πλήρω η ασυμμετρία τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε ένα μέλο το οποίο έχει του οικονομικέ, σε ένα μέρο το οποίο έχει στη διάθεσή του οικονομικού πόρου, από τη μία πλευρά και το μέρο εκείνο, το κράτο μέλο δηλαδή εκείνο από την άλλη πλευρά, το οποίο χρειάζεται, ε, έχει ανάγκη έκτακτη αυτούς τους πόρους. Άρα λοιπόν, αν λάβουμε υπόψη μα τα παραπάνω ε, και αν σκεφτούμε ποια είναι τα μέτρα τα οποία χρειάζονται ώστε να επανεξισορροπήσουμε την κοινωνική με την οικονομική διάσταση, ε, αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι οι μεταρρυθμίσει των συνθήκων, ώστε να υπάρχουν νέε κοινωνικέ αρμοδιότητε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αποτελούν προτεραιότητα. Αντιθέτω, δηλαδή, αυτό που συμβαίνει είναι οι νέοι μηχανισμοί διασφαλίζεται να είναι απλώ και μόνο ε, να συνάδουν με τι συνθήκε Ευρωπαϊκή Ένωση το χάρτη και ειδικότερα τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και στι διαδικασίε και επί τη ουσία. Πώ αυτό θα μπορούσε τώρα να επιτευχθεί όμω στην πράξη. Σε ό,τι αφορά τα πακέτα διάσωση, θα μπορούσαν λοιπόν αυτά να τεχθούν πλήρω υπό την, το πεδίο εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Για παράδειγμα, ε, ε, στην απόφαση Φλωρέσκου του 2017 το δικαστήριο βασίστηκε στο άρθρο 143 τη Εθνική Ελληνική τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε ό,τι αφορά την, ε, το πακέτο διάσωση για την Ρουμανία ε, και αποφάσισε ότι είναι αρμόδιο για να εκδικάζει ζητήματα συμβατότητα των μέτρων λιτότητα στη Ρουμανία αφενό και διατάξει ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα αφετέρου. Και γιατί εξέδωσε αυτή την απόφαση στο δικαστήριο, γιατί το μνημόνιο κατανόησης σύμφωνα με το δικαστήριο μπορεί να τύχει αναθεώρησης καθώς είναι δεσμευτικό και καθώ αποτελεί νομική πράξη ενό θεσμικού οργάνου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα συμπέρασμα το οποίο είναι εντελώ διαφορετικό από το συμπέρασμα που είχε φτάσει το δικαστήριο σε σχέση με αποφάσεις σε ό,τι αφορά άλλα πακέτα διάσωσης, όπως για παράδειγμα αυτό για την Κύπρο ή ε, το πακέτο διάσωση για την Ελλάδα ή ε, για την ε, Πορτογαλία. Άρα λοιπόν αυτή η δυνατότητα ex post εκ των υστέρων ελέγχου είναι πολύ ε, σημαντική, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι τα πακέτα διάσωση από τη στιγμή που ε, συντάσσονται συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και πώ μπορούμε να το εξασφαλίσουμε αυτό. Υπάρχει μια διάταξη στον ε, κανονισμό 472 του 2013, ειδικότερα το άρθρο 7 που ε, δεν λέει πολλά προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, απλώς αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη, εκείνο το κράτος μέλος που ζητά ε, οικονομική υποστήριξη, θα πρέπει να διαμορφώσει, να διατυπώσει ένα ε, πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, χωρίς να διευκρινίσει παραπάνω, ε, την πρακτική και τα, τα όσα ισχύουν εν είδη θεσμό σε ό,τι αφορά την, τον υπολογισμό των μισθών και το εθνικό πρόγραμμα αριθμαρίσης του κάθε κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 152 ε, τη Συνθήκη Λισαβόνα και το άρθρο 28 του Χάρτη. Κατά τη δική μου άποψη, θα πρέπει να γίνει μια αναδιατύπωση αυτού του κανονισμού που θα διευκρινίζει ότι αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να συνάδει με όλε τι κοινωνικέ διατάξει που περιλαμβάνονται στι συνθήκε και στο χάρτη. Επίσης αυτή η μετάλλαξη, αν θέλετε, η αναθεώρηση θα μπορούσε να ε, συμπεριληφθεί και στο πλαίσιο εκείνη της αξιολογήση αντικτύπου που είχε ε, υποστηρίξει ο πρόεδρος Γιούνκερ όταν είχε αναλάβει τα καθήκοντά της η σημερινή επιτροπή. Το πρόβλημα βέβαια ε, με τις αξιολογήσεις αντικτύπου είναι το πώς έχουν ε, χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, αν ρίξουμε μια ματιά στην αξιολόγηση αντικτύπου σε σχέση με το πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας ε, του 2015, ήταν μάλλον αστεία. Ήταν, γιατί ουσιαστικά αποτέλεσε ένα είδο συγνώμηση, ε, προσπαθούσε απλώ να δικαιολογήσει το γιατί ελαμβάνονταν τα σχετικά μέτρα και προβλέπουν αστικέ μεταρρυθμίσει ε, και δεν έκανε κάποια ε, κριτική εξέταση τη κοινωνική βιωσιμότητα αυτού του προγράμματο. Τώρα, εάν ρίξουμε μια ματιά γενικότερα στην οικονομική διακυβέρνηση και συγκεκριμένα στο εξάμεινο, έχουν γίνει κάποιε προσπάθειε σε ό,τι αφορά την το, την ενίσχυση τη κοινωνική διάστασης τόσο σε οργανωτικό όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο και υπάρχουν κάποια αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις περισσότερες για παράδειγμα συστάσεις οι οποίες υπάρχουν σε ό,τι αφορά όμως πάντοτε τη συμβολή τους για την επίτευξη των στόχων της Οικονομικής και Νομισματικής δηλαδή πάντοτε παραμένουν στον πυρήνα οι οικονομικοί στόχοι όχι οι κοινωνικοί και θεωρώ πως ε, ε, πραγματικά είναι αμφίβολο το ότι αυτές, αυτά τα πρώτα βήματα ε, αποτελούν ε, ουσιαστικά ένδειξη ότι θα σταματήσει να δίνεται προτεραιότητα στους οικονομικούς στόχους. Δηλαδή αυτές οι προσανατολισμένες προς την κοινωνική διάσταση συστάσεις έχουν οριακή σημασία σε σχέση με την παραδοσιακή εντός προσέγγιση και αυτό βέβαια δεν αποτελεί έγκληξη γιατί αυτό ε, εξάμεινο δημιουργήθηκε προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Κατά συνέπεια, λοιπόν, οποιαδήποτε κοινωνική στόχη είναι πάντοτε δευτερεύοντα σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, μπορεί κανεί να αναρωτηθεί ε, το κατά πόσο η υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων θα μπορούσε να, κάνει, να, να επιφέρει μια αλλαγή. Με βάση την ε, ετήσια έκθεση ανάδειξη του 2018, ε, βλέπουμε ότι η Επιτροπή αναφέρει ότι ο πυλώνας αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για την περαιτέρω εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και μια πηξίδα προκειμένου να υπάρξει περισσότερη σύγκληση ε, σε ό,τι αφορά τις καλύτερες ε, συνθήκες εργασίας και τις συνθήκες διαβίωσης. Και παρότι αυτό ακούγεται θετικό, μέχρι στιγμής ο πυλώνας έχει οδηγήσει μόνο στην ε, διατύπωση ε, ενός, μιας δέσμης δικτών που θα οδηγήσει στην καλύτερη παρακολούθηση ε, των, της επίδοσης των επιδόσεων των κρατών μελών σε σχέση με τα κοινωνικά ζητήματα. Βέβαια δεν θα ήταν δίκαιο το να κρίνουμε από τώρα το τι θα συμβεί σε σχέση με τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αλλά κατά τη δική μου άποψη θα χρειαστεί να γίνουν τεράστιες νομικές και πολιτικές προσπάθειες προκειμένου να ενεργοποιηθεί πραγματικά ένα τόσο αδύναμο εργαλείο όπως ο πυλώνας. Θα πρέπει λοιπόν να, γίνουν πιο, να ληφθούν πιο αποφασιστικά μέτρα ούτως ώστε ε, να λάβουν πιο σημαντικό ρόλο οι κοινωνικοί στόχοι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμενού. Και το έγγραφο εργασίας είναι αρκετά τολμηρό και συμφωνώ μαζί του γιατί ε, δείχνει να προτείνει ότι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη των κοινωνικών στόχων είναι ουσιαστικά η κατάργηση του εξαμήνου και εγκατάλειψη της, του βασι, της βασικής συλλογιστικής του εξαμήνου, ότι δηλαδή ε, η σύγκληση σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική αποτελεί απλώς και μόνο έναν τρόπο για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Και έρχομαι τώρα στα συμπεράσματα και, στην ολοκλήρωση της παρουσίασής μου. Ε, ο βασικός στόχος οποιασδήποτε μεταρρύθμισης ε, ε, με στόχο την ενίσχυση την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ε, κατευθύνεται πάντοτε προς την ενίσχυση του, του, του πολιτικού χώρου αν θέλετε των ε, περιθωρίων δηλαδή ελμών για να υπάρχει πραγματική κοινωνική πολιτική σε εθνικό επίπεδο. Και εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να γίνει εδώ μια αναδιανομή, αν θέλετε, τον, ανακατανομή των εξουσιών ανάμεσα στα υπερεθνικά θεσμικά όργανα αφενό και τα κράτη-μέλη αφετέρου. Όχι. Υπάρχει ήδη οικονομική και νομισματική ένωση και μια άλλη κατανομή των εξουσιών δεν θα λειτουργούσε αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή και μάλλον και για το ε, μέλλον που μπορούμε να προβλέψουμε, τα εθνικά κοινωνικά συστήματα θα αποτελούν τον πυρήνα ε, τον, ε, τον, τον ακρογωνίο λίθο της, της κοινωνικής διάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν αυτός ο στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί όχι μόνο με την εξορρόπηση μεταξύ οικονομικού και κοινωνικού σκέλους σε σχέση με τις διαφορετικές πολιτικές αλλά και με άλλα είδη δράσης. Για παράδειγμα, μέσω της δημιουργίας ε, ενός κεντρικού δημοσιονομικού μηχανισμού για την μεταφορά δημοσιονομικών κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελάντων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελέσει πράγματι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο. Γιατί τέτοιου είδου μεταβιβάσει μεταξύ των κρατών μελών θα μπορούσαν να μειώσουν τι πιέσει που ασκούνται στι κοινωνικέ πολιτικέ και θα μπορούσε να ξεφύγει από το ρόλο τη δηλαδή η κοινωνική πολιτική, το ρόλο που έχει σήμερα ω μεταβλητή δηλαδή προσαρμογή ε, ε, για του οικονομικού στόχου. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται ε, με πολλές ασάφειες και ανασφάλεια σε ό,τι αφορά τις ε, προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά τους τελευταίους μήνες. Τόσο σε ό,τι αφορά το ζήτημα της νομικής συμβάσης, όπως ανέφερε μόλις τώρα ο συνάδελφος, αλλά και σε ό,τι αφορά την ουσία. Γιατί ε, ακριβώς ένα ζήτημα ουσίας εδώ, το βασικό ζήτημα, είναι το κατά πόσο θα τεθούν προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά για την, την αυτών των κοντιλίων, το να τεθούν λοιπόν προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, μάλλον θα χρησιμοποιηθεί πολιτική με αιρεσιμότητες, δηλαδή επιβολή συγκεκριμένων υποχρεώσεων για την εκταμείωση των σχετικών ε, κοντιλίων. Και το δικαστήριο στην ε, περίφημη υπόθεση Πρέγκλ είχε ε, αποφασίσει ότι ο μόνος ο τρόπος ε, για να διασφαλιστεί η μεταβίβαση ε, τέτοιων κοντιλίων ε, προς ένα κάτω μέλος ε, δεν παραβιάζει την, τη σχετική ρήτρα μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εφόσον δεν οι προϋποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με μια τέτοια ε, ενίσχυση ε, δεν ε, οδηγούν στην επιβολή μιας ή μάλλον προωθούν την επιβολή μιας ορθής δημοσιονομικής πολιτικής. Άρα λοιπόν αυτή η ερμηνεία που έδωσε το δικαστήριο κατά δική μου άποψη χωράει αμφιβολίες γιατί ουσιαστικά ερμηνεύει με διαφορετικό τρόπο τη σχετική ρήτρα του no bailout, δηλαδή της μη ε, δυνατότητας μη εφαρμογή τη σχετική πολιτική εφόσον έχουν ληφθεί τα κονδύλια. Ε, παρόλα αυτά, μια τέτοια τοποθέτηση συνάδει και ε, με τις ε, ε, τοποθετήσει κρατών μελών όπως η Γερμανία και τα βόρεια κράτη-μέλη, ότι δηλαδή με, αυτές τις, ε, ε, με την επιβολή τέτοιων ρεσιμοτήτων ουσιαστικά θα μπορούσαν να μειωθούν οι ανησυχίες τέτοιων κρατών μελών. Εάν λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι τα ε, προγράμματα διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων συνάδουν πλήρω με τα όσα ε, προβλέπονται μέσα στη συνθήκη αλλά και στο χάρτη, ούτω ώστε να ξεφύγουμε από αυτέ τι ασφικτικέ ε, αιρεσιμότητε που τίθεται στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων διάσωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ευχαριστούμε για την ευκαιρία που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Συνοσπονδία των ε, Εργατικών Συνδικάτων να ακουστεί και να συμμετάσχει στην ε, συζήτησή σας. Έχουμε μια πλατφόρμα για το μέλλον της Ευρώπης. Τη λέμε για μια πιο ισχυρή Ευρώπη. Ευρώπης Δημοκρατικής και λοιπά. Και με αυτή η πλατφόρμα έχει αφετηρία το ότι θα πρέπει τα υψηλά, πρότυπα τα υψηλά στάνταρ, ε, τα βιωτικά, θα πρέπει να οδηγούν σε κάποια σύγκληση προς τα πάνω και για τους εργαζομένους να το πούμε ότι θα πρέπει αυτό να μεταφράζεται σε επαρκή κοινωνική πρόνοια, ε, δίκαιους ε, μισθού και συνδικές εργασία και μια αγορά εργασία που να διέπεται από κάποιου εκαθαρούς κανόνε και όλα αυτά στο άρθρο 3 το λέει η Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια κοινή αγορά και θα πρέπει να υπάρχει μια βιώσιμη ανάπτυξη με ισορροπία και ε, σταθερότητα τιμολογιακή, κοινωνική οικονομία της αγοράς και υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωση του περιβάλλοντος. Άρα, τι πήγε στραβά, αφού το Σύνταγμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση το προβλέπει όλα αυτά, γιατί όλα αυτά δεν μεταφράστηκαν σε πραγματικότητα και έτσι έχουμε τις ε, διεκδικήσεις των εργαζομένων. Οπότε θα πρέπει να σας ε, πω για κάποια πράγματα που έχουν συμβάλει ε, από πλευράς οικονομικής ε, στην αγορά και όχι από πλευράς κοινωνικής. Ε, πρώτα πρώτα έχουμε την ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ρωτήθηκε συγκεκριμένα το δικαστήριο ποια είναι η ορθότερη εφαρμογή της αρχής του δικαιώματος στην απεργία. Και, περίεργος, το δικαστήριο έκρινε ότι το δικαίωμα στην απεργία θα πρέπει να ασκείται αναλογικά και θα πρέπει η επίλυση του δικαιώματος να δικαιολογείται. Ε, αυτό είναι τελείως λάθος όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορώ να το κάθε νομικός. Γιατί θα πρέπει ο περιορισμός να δικαιολογείται. Ο περιορισμός να είναι ε, αναλογικός, όχι η άσκηση του δικαιώματος. Και αυτή η ιδέα, όπως είπε ο συνάδελφος, εδώ εξ αριστερών, ε, είναι, ότι εξηγεί πάρα πολλά η εν λόγω απόφαση του ΔΕΚ. Στη Συνδική της Λισαβόνας προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων ανθρώπων. Αυτό τι σημαίνει. Ότι στη συνέχεια οι έχοντες τα σχετικά δικαιώματα μπορούν να προσφύγουν στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να πει ότι πρόκειται εδώ για λάθος ερμηνεία του τι θα πει ανθρώπινο δικαίωμα. Αλλά περίεργος, παρά όλα αυτά τα οποία λέει η Συνδίκη της Λισαβόνας για τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι αυτά δεν συνάδουν προς την ε, συνθήκη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε σταμάτησαν όλα τα μέτρα, όλα τα διαβήματα για την προσχώρηση στην ε, ε, εν λόγω σύμβαση. Οπότε αν θέλουμε να λειτουργήσει το Σύνταγμα θα πρέπει να κάνουμε αυτά που λέει. Και το Σύνταγμα λέει ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στη Σύμβαση Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Δηλαδή ότι τα δεσμικά όργανα ε, θα πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και Ξέρω και το ότι θα πρέπει τα πράγματα να διορθωθούν. Ε, αλλιώς, δεν συνάδουν τόσο καν η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, αυτό δεν μπορεί να ισχύει αφού το λέει η συνθήκη θα πρέπει να το κάνουμε. Να προσχωρήσει στη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Ένωση. Άρα επίσης θα πρέπει να αναδειχθεί το θέμα του ότι κάτι πήγε στραβά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θέλουμε να έχουμε ένα πρωτόκολλο για την κοινωνική πρόοδο και το πρωτόκολλο το σχετικό θα πρέπει να τροποποιηθεί ούτως ώστε να ε, επιτρέπει να υπάρξουν οδηγίες για αντιστοίχηση των οικονομικών με τα κοινωνικά δικαιώματα. Να σας πω ακόμα δύο λόγια για το θέμα της ε, ε κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Είδαμε τι ε, επιφύλαξη έχουν οι καθηγητές για το ότι στο δίκαιο ακόμα αυτά ε, δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά. Θα πρέπει επίσης ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων να αναδειχθεί και βέβαια να αναγνωρίσουμε το, τη σκληρή προσπάθεια του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου ούτως ώστε να υπάρχουν δικαιότερες ε, συνθήκες και όροι εργασίας. Ε, οπότε έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Βέβαια, το θέμα είναι ότι τα, όλα αυτές τις προσπάθειες προσκρούν στα κράτη-μέλη και είχαμε τα όσα εξήγηλε νωρίτερα φέτος ο πρόεδρος Γιούνκερ, ούτω ώστε να έχουμε ειδική πλειοψηφία σε κάποιες αποφάσεις ε, σχετικές με αυτά τα ζητήματα. Ούτε ισχύει ότι τα μέτρα για να είναι δικαιότερη αγορά θα μπορούν να φρενάρουν ε, με βέτο ενός κράτους μέλους. Πρόοδος θα ήταν εάν δεν υπήρχε τέτοια, τέτοια προϋπόθεση, τέτοια πρόβλεψη αυτού του βέτα λοιπόν που φρενάρει την πρόοδο. Τώρα όσον αφορά ε, το, το, το, πόσο αφορ, το πόσο ωφελεί ο πυλώνας αυτός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε σύσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και υπάρχει κάποια πρόταση σε σχέση με ε, κάποιο είδους ε, στόχο ε, οπότε για αυτό το λόγο ε, θα πρέπει να γίνουν κάποιες περικοπές ε, αυτό όμως θα πρέπει να, να εξεταστεί για το αν εμπίπτει στον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα μπορούσε επομένω να είναι κάτι σαν ασπίδα αυτός ο πυλώνας ότι τα κράτη-μιλή δηλαδή τηρούν τις υποχρεώσει τους για αυτά τα κοινωνικά δικαιώματα. Να, εδώ είναι ένας τομέας που επιβάλλει να τροποποιηθεί η συνθήκη. Και αυτό πρέπει να συζητηθεί με τους Ευρωπαίους. Θέλετε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο δραστήρια υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ή μήπως θεωρείτε ότι καλύπτεται αυτή η προσπάθεια ήδη από τόσο κάνουμε. Πώς θα γίνει να εργαστούν τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει δηλαδή ότι είναι περισσότερο ασπίδα αλλά όχι ξύφος ε, ο πυλώνας αυτός. Επίσης έχουμε κάποιες διατάξεις στο Σύνταγμα που αφορούν τους κοινωνικούς εταίρους. Μας προβληματίζει το εξής. Η Επιτροπή δεν κάνει αυτό το οποίο πρέπει όσον αφορά την ε, νομοθεσία ε, η οποία θα πρέπει να είναι δεσμευτική, να είναι πιστική για τους ε, εργοδότες αλλά και για τους εργαζομένους. Έχει αρνηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυθυγραμμίσει την νομοθεσία της με την συνθήκη και έχουμε ήδη τώρα μια υπόθεση σχετική που βρίσκεται ενώπιον του εισαγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπότε και εδώ χρειάζεται μια τροποποίηση της συνθήκη, ή τέλο πάντων να κατανοηθεί το τι λέει η συνθήκη. Διότι και εργοδότες και εργαζόμενοι πρέπει να προτείνουν το πώς θα λειτουργούν τα νομοθετήματα. αν το δικαστήριο καταλήξει ότι δεν λειτουργεί έτσι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα ήταν ε, τρομερό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα είχε με πολύ μεγάλη σημασία αν ε, γίνονταν, αν είχαμε τέτοιου είδου ε, απόφαση που θα ήταν πάρα πολύ σημαντική και για εργαζόμενους και για εργοδότες. Μα ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι το Σύνταγμα. Εγώ τους λέω ότι είναι οι πιο βασικοί κανόνες που διέπουν ας πούμε ένα σπίτι ε, ότι καθορίζει το πώς μπορούμε να συνεπάρξουμε. Και το ίδιο αφορά και το Δινές Γραφείο Εργασίας τοποθετήθηκε για όλα αυτά που συζητούμε τις τελευταίες εβδομάδες τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και λέει ότι παγκόσμια ειρήνη μπορεί να υπάρχει μόνο όταν βασίζεται σε κοινωνική δικαιοσύνη. Πριν από 100 χρόνια. Ίσχυε αυτό. Την εποχή του Παγκόσμιου Πολέμου και ισχύει και τώρα. Και αυτό είναι το μήνυμα των εργαζομένων. Ότι χρειάζεται ειρήνη, χρειάζεται κοινωνική δικαιοσύνη και αυτά θα πρέπει να μπουν να κατοχυρωθούν στο σώμα της ε, συνθήκης και να πετύχουμε σε αυτό το μέτωπο όπως πετύχαμε στο μέτωπο της οικονομίας. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Έχουμε άλλα 25 λεπτά. Για ερωταπαντήσεις. Κάντε ό,τι μπορείτε συνάδελφοι τώρα που έχουμε εδώ τους ειδικούς καλεσμένους μας. Ε, βέβαια, και ο Φα... έφυγε ο Φάμπιο. Ε, μόνο η Μπάρμπαρα έχει μείνει. Ε, η Μπάρμπαρα είναι επίσης ε, μία εμπειρογνώμονα και μπορούν να μιλήσουν και όποιοι θέλουν εκ των σχεδόν εισηγητών. Και εσεί. ναι. Μπάρμπαρα, σύντομα, 5 με 7 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ε, τρεις ομιλητές. Είναι πολύ σημαντικά τα όσα συνέβαλαν στη συζήτηση. Και όλα αυτά θα, θα αποτελέσουν προσθήκη στο έγγραφο εργασία μας. Είπαμε για τους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους πατέρες της Ένωσης, που το θυμάμαι ότι ε, είχαν το κοινωνικό ιδεώδες ε, υπόψη τους. Το είχαν ενστερνιστεί και συγκεκριμένα αναφέρομαι στο beverage όσον αφορά την, ε, ε, το γενικό ιδεώδες τέλος πάντων και για την εγγύηση κάποιου εισοδήματος για τους μη προνομιούχους. Επίσης, με την ευκαιρία για να δούμε κάποια ζητήματα του εγγράφου εργασίας που ετοίμασα με τον Φάμπιο Μάσιμο Καστάλτο. Εμείς είχαμε ως ε, αφετηρία μία ε, διαπίστωση ότι από πλευράς κοινωνικής Οικονομική και Νομισματική Ένωση κατά κάποιο τρόπο απέτυχε, δεν είναι βιώσιμη και ως αφετηρία μας λοιπόν είχαμε ότι υπάρχει πάρα πολύ κοινωνική ισορροπία, ανισορροπία, συγγνώμη, και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο από την δημοσιονομική έλλειψη ισορροπίας. Οπότε παρακαλώ να μας πούν τη γνώμη τους επ' αυτού οι καλεσμένοι μας. Τι γνώμη έχουν για τις προστριβές, τις διαπραγματεύσεις, ας πούμε, μεταξύ Ένωσης και Ιταλικής κυβέρνησης. Μα οι ευρωπαϊκές αρχές δεν έχουν λάβει καθόλου υπόψη το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση στην Ιταλική κοινωνία και ότι έχουμε 6 εκατομμύρια ε, ατόμων που βρίσκονται σε απόλυτη φτώχεια. Μα τι θα γίνει, τι προϋπολογισμό να κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά την στρατηγική για το 2020 και αυτή θεωρούμε ότι έχει αποτύχει. Ε, είδαμε τι γίνεται με τα 20 εκατομμύρια των φτωχών και να μην αλλώσω όλο το χρόνο αλλά είπαμε στο έγγραφο εργασία μας ως πρόταση το εξή. ότι θα πρέπει να ισχύσει, να τηρηθεί ο κοινωνικός χάρτες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα πρέπει τα τις κοινωνικές πολιτικές να μπουν στην ε, συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η εγκατάλειψη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τέλος πάντων η εκβάθρον αναθεώρησή του θα πρέπει να ισχύσει. <coughs> και έτσι οι κοινωνικές παράμετροι να αποκτήσουν προτεραιότητα. Και κάτι να γίνει με το ελάχιστο εισόδημα. Να πολλά πολλά μπορούσαμε να προσθέσουμε, αλλά τέλος πάντων όσον αφορά την τροποποίηση της συνθήκης έχω να πω ότι κατά τη γνώμη μου πολλά πολλά θα μπορούσαν να γίνουν, πολλά μπορούσαν να αλλάξουν στην ισχύουσα συμφωνία. Καλά έχουμε το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Σήμερα η Επιτροπή δεν το έκρινε. Αλλά πάντως περιέχονται πάρα πολλά στοιχεία για την συνθήκη. Ένα κοινωνικό πρωτόκολλο δεσμευτικό. Όχι, όχι ο κοινωνικός πυλώνας του Γιούγκερ. Ε, αυτό είναι τίποτα, είναι κάτι χωρίς περιεχόμενο. Σαν ένα μύδι, ένα στρίδι τροφό που δεν έχει τίποτα μέσα. Ε, η τήρηση του εξαρτάται μόνο από την καλή πίστη. Πολλά πολλά θα μπορούσα να πω, αλλά θα βάλω τελεία εδώ. Και γι' αυτό σας. Ε, σας παρακαλώ αν μπορείτε συσχετίστε αυτά τα οποία μας λέτε με τη δουλειά μας. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για αυτές τις τρεις παρουσιάσεις. Μας έδωσαν πολύ σημαντικά ερεθίσματα για σκέψη. Ο πρόεδρος Ζούκερ είχε αναφέρει όταν είχε αναλάβει τα καθήκοντά του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει ένα τριπλό α ως βαθμολογία σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάσταση. Και συμφωνώ μαζί σας ότι παρασάγκα απέχομαι από ένα τριπλό α. Ε, αντιθέτως η ψαλίδα εντός εισαγωγικών ανάμεσα σε φτωχού και πλουσίους στα κράτη-μέλη έχει ανοίξει ακόμα περισσότερο, έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Ε, στο πλαίσιο λοιπόν τη επόμενης βουλευτική ε, ε, η κοινωνική διάσταση θα πρέπει πραγματικά να αποτελέσει προτεραιότητα. Καθώς βρισκόμαστε υπό πίεση χρόνου, να πω πως ε, συχνά ε, σωστά αναφέρατε ότι οι κίνδυνοι στα διαφορετικά κράτη-μέλη ή σε ορισμένα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να αποτελέσουν κινδύνου γενικευμένου για όλα τα κράτη-μέλη, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε κοινού σταθεροποιητέ. Και αυτό ισχύει. Δηλαδή είμαστε μια ένωση πραγματική και υπάρχουν δηλαδή στοιχεία και οικονομικά και δημοσιονομικά μεν, αλλά και κοινωνικά στοιχεία και κοινωνικοί σταθεροποιητέ που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Ίσως ε, θα μπορούσαμε ε, να προβλέψουμε ένα είδος νομοθεσίας ή νόμου σύγκλησης, στον οποίο λοιπόν νόμο αυτών σύγκλησης θα μπορούσαμε να αναφέρουμε με βάση και την ε, οικονομική ισχύ κάθε κράτους μέλους ποιε είναι οι δαπάνες σε ό,τι αφορά το τομέα της παιδείας, ποιε είναι οι δαπάνες σε ό,τι αφορά το κοινωνικό σύστημα και ό,τι καθεξής, έτσι ώστε πάντοτε να γίνεται μια αναβάθμιση, δηλαδή προς τα πάνω, μια αύξηση ε, και όχι μείωση. Γι' αυτό σας ε, το θέτω το ερώτημα και σε σχέση με το ευρωπαϊκό εξάμεινο το οποίο ετέθη μόλις τώρα. Αυτά τα ερωτήματα τα ε, έθεσα στον πρώτο μελετή, τώρα στον ε, κύριο Κασταμάνια. Αναφερθήκατε στο ότι θα μπορούσαμε σε ό,τι αφορά τα προγράμματα διάσωσης να προβλέψουμε ε, την ένταξη νομοθεσία, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το, ε, τη ρήτρα Out. Ε, Και βέβαια αυτό ισχύει ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις μεταβιβάσεις και το γεγονός ότι έχουμε τα ισχυρά κράτη-μέλη τα οποία ενισχύονται ακόμα περισσότερο και τα δύναμα κράτη-μέλη που εξασθενούν ε, ακόμα περισσότερο. Άρα αυτό που χρειάζεται πράγματι είναι ότι χρειάζονται μεταβιβάσει σε ό,τι αφορά συγκεκριμένους τομείς, όπως είπε και άλλοι. Άρα λοιπόν, ρωτώ, ε, κύριε Κωνσταντινίδη, μήπω ε, θα μπορούσαμε να έχουμε μεταβιβάσει τέτοιου είδου δημοσιονομικέ σε ό,τι αφορά συγκεκριμένου τομεί και όχι γενικέ μεταβιβάσει. Αυτά λοιπόν προ τον κύριο Κωνσταντινίδη. και τώρα πεσυνόμενο τη κυρία Έστρε Λίντ. Να πω ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε εδώ να αναλάβει δράση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Δικαστήριο. Ε, γιατί αυτό θα διαρκέσει πολύ και ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας και τις τοποθετήσεις του Δικαστηρίου. Άρα λοιπόν χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι δεν ε, τυχάνουν ε, δευτερεύουσα αν θέλετε μεταχείριση ή κοινωνική στόχοι σε σύγκριση με του οικονομικού ε, στόχου. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τέτοιο project αφού κατοχυρώνονται και τα κοινωνικά ε, αυτά ζητήματα στη συνθήκη. Με άλλα λόγια, αυτό που λέω είναι ότι ενδεχομένως θα καταστεί απαραίτητη η αναδιατύπωση της συνθήκης. You didn't uh, ήθελες να πάρει το λόγο ή όχι. Ραμόν και μετά εσύ Μεσέντες, στο συγγνώμη γιατί έκανα κάποιο λάθος. Grazie, ma non era, non era necessario. Α, καλά, καλά, μια που μιλάει ο Ραμόν στο τηλέφωνο, να σας τα πω. Ε, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κινηθούμε σε δύο επίπεδα. Πρώτο πρώτο. Αυτό που συζητούμε σήμερα και από την άλλη μεριά είναι το θέμα του κοινωνικού πυλώνα που θα πρέπει ίσως να αναθεωρηθεί, να απλουστευτεί και να μπει στη συνθήκη. Ε, χάθηκε η μάχη για να μπουν τα κοινωνικά στη συνθήκη και τέλος πάντων εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική ο κόσμο αγώνας για να γίνει στο μέλλον μια αναθεώρηση της συνθήκης. Τώρα, όσον αφορά την ε, νομοθεσία την κοινή μη συνταγματική νομοθεσία. Μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Σήμερα η πολιτική μας ομάδα κατέβασε την ε, πρόταση για αλλαγή του ευρωπαϊκού εξαμήνου και του τρόπου διαχείρισης του. Αν εμείς μπορούσαμε ε, αυτά που λέτε, αυτά που λένε τα συνδικάτα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, όχι μόνο τις οικονομικέ μεταβλητές, αλλά και κοινωνικές ε, και περιβαλλοντικές μεταβλητές. Στόχους δηλαδή που θα πρέπει να επιτευχθούν και από τα κράτη ξεχωριστά. αλλά και για το περιβάλλον. Αν θέλουμε να είμαστε βιώσιμοι ως ε, κοινωνία, άρα θα πρέπει όλα αυτά, οι στόχοι δηλαδή περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία, όλα αυτά να αποτελέσουν ε, ένα, ένα σύνολο, μια σύγκληση ε, στόχων που πρέπει να είναι συμβιβατοί μεταξύ τους. Αυτό θα πει συνοχή. Και σε σχέση με, το, με στόχους του 2020 για την Ευρώπη επίσης. Δεν θα πρέπει να έχουμε απόκληση αλλού να πηγαίνει ο ένας στόχος και αλλού να πηγαίνει ο άλλος. Επομένως ε, είναι αναγκαίο να υπάρχει σύγκληση. Οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον. Απαραίτητα αυτά. Και έτσι θα έχουμε βιωσιμότητα πολιτικών, μακροπρόθεσμη. Πέστε μας, τι πιστεύετε για αυτά τα δύο επίπεδα. Αφενός το πώς θα κινηθούμε κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και έτσι να υπάρξει μια καινούργια ερμηνεία, καινούργια σύλληψη για την βιωσιμότητα σε κάθε χώρα. Και από την μεριά να μπουν συνθήκε. στόχοι και αυτό εννοούσε ο, ο Γιούνκερ όταν μίλαγε για τον κοινωνικό πυλώνα. Άρα και στις κατευθύνσεις να υπάρξει αυτός ο στόχος της βιωσιμότητας και αυτοί οι στόχοι να ληφθούν υπόψη παντού και όχι μόνο δημιουργικά. Εκεί να κατατείνουν οι προσπάθειες για το πώς η τροποποίηση των συνθήκων θα αποτελέσει ε, μια άλλη, θα δώσει μια άλλη μορφή στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Δύο λεπτά στο Ραμόν και στον Χέλμουτ, γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι εμπειρογνώμονες. Ναι, μάλιστα δεν έχω πρόβλημα. Δύο λεπτά. Ε, Άκουσα την κυρία Λίντς που μας μίλησε για την σημασία του να προσχωρήσει η Ευρώπη στην Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ακριβώς όπως ορίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Και έμεσα επικρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ότι δεν γίνεται μια τέτοια κίνηση. Όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια γνωμοδότηση που αποσκοπεί στο να ρυθμίσει τα της προσ... προσχώρησης της Ένωσης στην Σύμβαση. Όμως από το δικαστήριο υπήρξαν πάρα πολλές ενστάσεις που ακόμα τις συζητάμε. Άρα είναι άδικο να αποδίδεται ε, έλλειψη βούλησης ε, ή αμέλεια στο κοινοβούλιο. Γιατί κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, απλώς περιμένουμε από τεχνικής πλευράς να λυθούν οι έξι, αν δεν κάνω ενστάσεις του 10. Χέλμουντ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν. Και είναι σημαντικό να υπάρχει ένας ε, ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων. Μεταξύ ημών εδώ στην αίθουσα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όμως το ζήτημα είναι ότι δεν συνδέουμε αυτή την πρόκληση με όλες ε, τις ε, εκθέσεις που εκπονούμε εδώ και χρόνια. Για το μέλλον της Ευρώπης, για την Τραπεζική Ένωση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά συνδέονται με το ζήτημα του κοινωνικού πυλώνα και κατά πόσο τον ενσωματώνουμε σε όλη την ομαθητική μας δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ας πούμε, τα όλα αυτά, εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σας ε, ρωτώ ποιους τρόπους διαβλέπετε εσείς για να αλλάξουμε τη στάση του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς αυτήν την κατεύθυνση. Διαφορετικά, ό,τι και να λέμε εμείς για την κοινωνική διάσταση, δεν μας πιστεύει ο κόσμος. Γιατί η εμπειρία στην καθημερινή μας ζωή είναι τελείως αντίθετη από αυτό που συζητούμε εδώ. Και ο Ραμόν πολύ σωστά λέει ότι δεν είναι θέμα του Κοινοβουλίου γιατί δεν έχουμε εμεί το δικαίωμα πρωτοβουλία νομοθετική. Πώ μπορούμε λοιπόν να αυξήσουμε τη συνείδηση του κοινού ότι είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη της Ένωσης. Εγώ εδώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου ή μάλλον εγώ είμαι εδώ Αυστηρή, με το ρολόι. Θα σας δώσω λοιπόν τρία λεπτά. Έχουμε και ένα κείμενο της κυρίας Λίντς που μας είπε ότι θα το στείλει. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, τρία λεπτά έκαστος. Ευχαριστώ πράγματι πολύ σημαντικά τα σχόλιά σας. να σχολιάσω αυτά που είπατε για τον κοινωνικό πυλώνα. Η κυρία Σπινέλη είπε ότι ο κοινωνικός ε, πυλώνας είναι μόνο στα λόγια. Εγώ θα ήθελα να είμαι λίγο πιο επικαδηματικός. Είναι θετική η εξέλιξη ο κοινωνικός πυλώνας, γιατί τουλάχιστον υπάρχει μία Ενεολογική συμφωνία και συνοχή. Το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ συνάδει με ε, τις αρχές της ε, κοινωνικής, ε, του κοινωνικού πυλώνα. Και αυτό από μόνο του έχει μια αξία. Από εκεί και πέρα έχετε δίκιο. Αν δεν δώσουμε αυτά αποτελέσματα, θα μας γυρίσει μπούμεραγκ. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αποτελέσματα. Όμως δεν νομίζω ότι εδώ πρέπει να μετατρέψουμε και τις 20 ε, αρχές ε, σε νομοθετικές, δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις. Είναι προβολικό. Θέλουμε όμως έναν ε, οδικό χάρτη, κάτι που μας λείπει, ούτω ώστε κάποιες από τις αρχές να περάσουν στην νομοθετική διαδικασία, άλλες Ε, να αποτελούν οδηγό για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Άλλες αρχές θα πρέπει ε, να συμβάλλουν στην καθοδήγηση των ε, χρηματοδοτικών μηχανισμών που έχουμε και που θα αναπτυχθούν και στο μέλλον από πρακτική άποψη. Να σα δώσω αρχικά ένα θετικό παράδειγμα. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για την επανεξέταση της οδηγίας γραπτής αναφοράς που είναι πολύ σημαντικό γιατί αφορά την ποιότητα και την προβλεψιμότητα της εργασίας μας και εκεί χρειαζόμαστε πραγματικά δεσμευτική νομοθεσία. Ένα άλλο παράδειγμα που δεν είναι τόσο θετικό και με προβληματίζει. Βασικό στοιχείο ήταν η διασφαλισμένη πρόσβαση στην ε, κοινωνική προστασία. Όποιος εργάζεται λοιπόν θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε επαρκή κοινωνική προστασία αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει ότι θα υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία και σιγά σιγά διολυστήσαμε προς ε, μία ανακοίνωση. Και για πολιτικούς λόγους έγινε αυτό. Σύσταση μάλλον όχι ανακοίνωση. Έχουν λοιπόν μία πιο ήπια προσέγγιση τώρα, ένα βήμα προς τα πίσω, μια παναχώρηση και τώρα πρέπει να αδράξουμε αυτή την σύσταση και να σημειώσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη πρόοδο. Στα κράτη-μέλη λοιπόν υπάρχει πρόσβαση σε όλους ε, όσοι εργάζονται στην κοινωνική προστασία. Λοιπόν, κλείνοντας, δεν είμαι αρνητικό συνολικά. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει ε, λήξει το ζήτημα. Υπάρχει ένας κίνδυνος αν ε, δεν τα μετατρέψουμε όλα αυτά σε αυτά τα αποτελέσματα μπορεί όντω να λειτουργήσει εναντίον μα. Δεν χρειάζεται όλα αυτά να γίνουν ε, δεσμευτική νομοθεσία. Κάποιες αρχές ναι, άλλες όχι. Άλλες αφορούν την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και για άλλες αρχές ε, το κρίσιμο στοιχείο είναι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δυόμιση λεπτά για τους άλλους δύο. Λοιπόν, δεν έχω πολύ χρόνο, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματά σας, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, πρώτα, κατά πόσο το Ταμείο Συνεχής μπορεί να ε, θεωρηθεί, να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά προς ε, την μεταφορά. Ναι, και στο πλαίσιο της αρεσιμότητας και στο Ταμείο Συνοχή έχουμε το ίδιο πρόβλημα, ότι μπορεί να έχουμε το ίδιο πρόβλημα που είχαμε και με τα πακέτα διάσωση. Πρέπει να το αποφύγουμε αυτό, κατά τη γνώμη μου. Μετά, δεν ξεχνώ και την συμβολική αξία αυτών των μεταφορών, γιατί δημιουργούν και μια αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, δεν έχουν ακριβώ την ίδια διάσταση. Το ερώτημα της κυρίας Μπρέσο για ε, ριζική αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμφωνώ απολύτω, θα ήταν κάτι πολύ θετικό, όμως οι κυρώσει ε, που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ασκήσει πίεση στα κράτη-μέλη συνδέονται ακόμα με οικονομικά και νομισματικά ζητήματα. Καλές οι συστάσει, λοιπόν, αλλά κάποια στιγμή, όταν δυσκολέψει το πράγμα, έχουμε τις πραγματικές κυρώσεις. Οπότε είναι δύσκολο να τα συγκεράσουμε. Και τέλος, τι πρέπει να κάνουμε. Ως νομικός ντρέπαμε που το λέω, αλλά βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον νόμο, ενώ η πολιτική είναι αυτή που θα πρέπει να σημειώσουν το επόμενο βήμα. Έχουμε πολύ καλά ε, νομικά εργαλεία αυτή τη στιγμή το ευρωπαϊκό σταγματικό πλαίσιο είναι ουδέτερο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε. Ελπίζουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές και να έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μεγαλύτερο, πιο έντονο κοινωνικό προσανατολισμό και να αξιοποιήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σε ένα πνεύμα που ευθυγραμμίζεται περισσότερο με το πνεύμα των εθνικών φυσικά ως νομικός θεωρώ ότι το νομικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά δεν μπορεί να τα λύσει όλα από μόνο του. Η πολιτική συνένεση λοιπόν θα πρέπει να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Διαφορετικά, είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε το παραμικρό και κοινωνικό πρωτόκολλο μπορούμε να έχουμε και ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά χωρίς αυτό δεν υπάρχει πρόοδο. Ευχαριστούμε κυρία Λίντ. Ευχαριστώ. Φυσικά και δεν ήθελα ε, να σας επικρίνω, να επικρίνω το Κοινοβούλιο, αλλά να σας ενθαρρύνω. Εφιστά την προσοχή σας όμως στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λέει ότι ε, η προσχώρηση ε, ε, εκρεμεί και είναι το δικαστήριο που ε, παρεμποδίζει τη δικασία και μετά αναφέρεται ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί αυτό να επιληθεί. Είναι όμως τρομακτικό κάτι τέτοιο, γιατί αν δεν κάνει αυτό που πρέπει, δηλαδή να διορθώσει τα κακό κείμενα, τότε ο κόσμος, ο κόσμος θα αρχίσει να χάνει την εμπιστοσύνη του, την πίστη του, ευρύτερα στο πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σημειώστε λοιπόν ότι εγώ ε, αναφέρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ε, βασικό ομοχλό ε, προώθησης του αιτήματο προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Για το κοινωνικό πρωτόκολλο σίγουρα είναι μια ιδέα που έχει οριμάσει και ελπίζουμε στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υπάρχει μια κατανόηση για το πόσο σημαντικό είναι να διορθώσουμε εδώ την ε, συνθήκη, αλλά και θα εντοπίσουν τι μπορεί να γίνει στο πλαίσιο των διατάξεων. Με ρωτήσατε τι μπορούμε να εξετάσουμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ένας ελάχιστος ε, μισθός στην Ένωση θα μπορούσε να είναι το 60% του μέσου ή του εθνικού. Θα μπορούσαμε επίσης να έχουμε περισσότερες ε, συλλογικές ε, διαπραγματεύσεις για να υπάρξει μια εξισορρόπηση της κατάστασης στην αγορά εργασία. Γιατί πολλές επιχειρήσεις πραγματικά ε, σαρώνουν την αγορά εργασίας, ε, εκμεταλλεύονται στο έπακρο τη σημερινή ε, αστάθεια. Πρέπει να δώσουμε περισσότερη δύναμη στους εργαζομένους να συμμετέχουν σε συλλογικέ διαπραγματεύσεις να πάρουν το μερίδιο που του αναλογεί και να διορθωθεί η κατάσταση στην εσωτερική αγορά η ενωσιακή συνθήκη, θα μου πείτε, δεν μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό. Δύο στοιχεία. Πρώτον, υπό το εξάμεινο δεν εμπόδισε όμως ε, την ΕΚΤ και άλλα θεσμικά όργανα να ε, δώσουν συστάσεις για την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σε, σε κλαδικές διαπραγματεύσεις μάλλον. Επομένως, με ποιο επιχείρημα μπορείτε να μου πείτε ότι αυτό δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε και σε άλλες ε, περιστάσεις. Δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία αυτού του επιχειρήματος στους εργαζομένους. Σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δώσατε και πράγματι θα στείλουμε λεπτομερή παρέμβαση και για το κοινωνικό πρωτόκολλο. Σας ευχαριστώ πολύ ξενόματος της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι πάντα μια δύσκολη συζήτηση και νομίζω ότι μας έχετε δώσει και παρουσιάσει και νέες διαστάσεις. Μου άρεσε πολύ η τοποθέτησή σας ως νομικού ότι πρέπει ε, να προωθήσουμε και τις νομοθετικές και τις πολιτικές αλλαγές. Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε και τα κείμενά σας. Ε,